δημοσιεύτηκε η αυριανή ημερήσια διάταξη για την Ολομέλεια. Σας εύχομαι και σας κύριε Επίτροπε στις ε, υπαλλήλους, στους συναδέλφους και σε, στις δικούς μας υπαλλήλους και στους διερμηνείς καλή ανάπαυση πέρα στη συνεδρία σας.